Uh, Mr. good morning. We can... Αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα. Ας ξεκινήσουμε με την ε, ψηφοφορία. Είμαστε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχει εγκριθεί. Λοιπόν, ψηφίζουμε για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα. Ελπίζω να έχετε τις ε, κάρτες σας. Λοιπόν, ξεκινάμε. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 4 με την προφορική τροπολογία κυρία Ροζιέρ προφορική τροπολογία ε, θέλω να υποβάλω εξ τις της ε, κυρία Βιόλ που δεν, ήταν εδώ, που δεν μπόρεσε να είναι εδώ σήμερα. Θέλω να σας το διαβάσω λοιπόν. Στο τέλος του συμβαστικού κειμένου η, τροπο, η προφορική τροπολογία διευκρινίζει την αναφορά στα προαναφερθέντα έγγραφα και υπογραμμίζει την όρους agenda και meetings. Δηλαδή λέει, είναι της άποψης ότι ο κατάλογος τριμερών ε, συναντήσεων και η ατζέντα τους, θα πρέπει, η μερίσια τους διάταξη θα πρέπει να γίνεται άμεσα διαθέσιμη στο Κοινοβούλιο. Και μετά το υπόλοιπο συνεχίζει το ίδιο. Κυρία Χάουταλα. Εγώ Σας ευχαριστώ. Την ε, στηρίζω και να εξηγήσω γιατί Νομίζω πως καταλήξαμε σε μια ευρύτατη συμφωνία για να αυξηθεί η διαφάνεια και η πρόσβαση στα έγγραφα και στα μήτρώα του Κοινοβουλίου για κάποια έγγραφα τριμερών διαλόγων. Αλλά υπάρχει ένα θέμα που ακόμα θα συζητηθεί στο μέλλον. Δεν συμφωνήσαμε από αυτού και ίσως ε, λυθεί από μια υπόθεση που εκρεμεί στο δικαστήριο και αφορά τα λεγόμενα έγγραφα της τέταρτης ε, στο πλαίσιο του τριμερούς διαλόγου. Νομίζω λοιπόν πως η συμφωνία που έχουμε μεταξύ όλων των ομάδων είναι πολύτιμη και θα προχωρήσει την ε, συζήτηση. Ε, thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οπότε ψηφίζουμε. Η γραμματεία με ενημερώνει πως υπάρχουν δύο σοσιαλιστές, ένας σοσιαλιστής ε, που δεν μας έχει κοινοποιηθεί γραπτός εκ των προτέρων. Okay, okay, Ωραία, μάλιστα. It seems to be fixed, however, uh, may inform the political group. εντάξει. Ε, ορθώθηκε. Εάν τα μέλη που δεν είναι τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής έρχονται στην ψηφοφορία πρέπει να ενημερώνεται η γραμματεία ε, εκ των πρότερων. Λοιπόν, συμβαστική 4 υπέρ. Με την προφορική τροπολογία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 Τροπολογία 15. Απορρίπτεται λοιπόν. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική ψηφοφορία ψηφίσματος. Εγκρίνεται συγχαρητήρια στην κυρία Χάουταλα. Now we continue. Συνεχίζουμε και κλεισμένων των θυρών.